και σε μια μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα τη συζήτηση. Και τώρα, βάσει της ημερήσιας διάταξης, φτάνουμε στη δήλωση τη Αντιπροέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη είπα τη εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, για την ε, πολιτική για την περιοχή της Αρκτικής. Εξ ονόματος της Αντιπροέδρου, ο Επίτροπος Φούλη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναβαθμίζει τη συνεισφορά τη ε, στην αρκτική συνεργασία και γι' αυτό με τα χαράς βρίσκομαι εδώ να μιλήσω στο Κοινοβούλιο εξ ονόματο της ε, υπάτης εκπροσώπου της κυρίας Άστον για την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωση για την Αρκτική μετά από την έγκριση της κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη υπάτης εκπροσώπου τον Ιούνιο. Έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ε, γίναμε ο μεγαλύτερος χορηγός ε, της έρευνας στην Αρκτική με συνεισφορά της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επιπλέον, ο τμήμα της ε, περιφερειακής και διασυνοριακής χρηματοδότησής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τοποθετήσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε οικονομική ανάπτυξη από τη Γρυλανδία μέχρι τη Ρωσία αν ε, προσθέσουμε σε αυτά και την ε, διμερή συνεισφορά των κρατών μελών και φτάνουμε πλέον σε ένα ποσό περίπου 2 δισεκατομμύριων ευρώ. Τα επόμενα βήματα τα οποία σχεδιάζουμε θα οδηγήσουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρκτική συνεργασία σε πιο ουσιαστικά στοιχεία. Η πολιτική μας εδράζεται σε τρεις βασικές πτυχές. Γνώση, ευθύνη και δέσμευση. Ξεκινούμε με τη γνώση. Ο νέος ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα δημιουργήσει στενότερους δεσμούς με τους ερευνητές από τρίτες χώρες. Εξετάζουμε επίσης κατά πόσον θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ενημέρωσης για την Αρκτική. Να περάσουμε τώρα στην ευθύνη. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας ε, στην Αρκτική και με τον ιδιωτικό τομέα για να αναπτύξουμε ε, τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον χαμηλού κινδύνου που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν εξορρεκτικές βιομηχανίες και ε, η ναυτιλία. Και τέλος, όσον αφορά τη δέσμευση, ενισχύουμε τον διάλογό μας με όλες τις χώρες της Αρκτικής και όλους τους ενδιαφερομένους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να δεσμεύεται με τις αυτόχθονες ομάδες της Αρκτικής για να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε σε αρκετούς πρακτικούς τομείς. Θα οργανώσουμε ένα διάλογο αυτοχθόνων στη, ε, της Αρκτικής στους επόμενους μήνες. Και ε, είμαστε και να αναμονή τη σημαντική απόφαση για το καθεστώ παρατηρητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από τα οκτώ ε, κράτη της Αρκτικής που αποτελούν το Αρκτικό Συμβούλιο και κατά την άποψή μας είναι και το βασικό διεθνές φόρουμ που ασχολείται με θέματα της Αρκτικής. Είμαστε βέβαιοι ότι τα μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου θα καταλήξουν σε μια δίκαιη απόφαση, θα αναγνωρίσουν την πολύ σημαντική συνεισφορά που μπορεί να ε, επιφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο έργο του Αρκτικού Συμβουλίου και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να βοηθήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του που προέρχεται από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ολοκληρώνοντα να σα πω ότι οτιδήποτε και αν κάνουμε, ένα πράγμα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει για την Αρκτική. Και αυτό είναι να συνεργαστούμε με του διεθνεί εταίρου μα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα τη αλλαγή του κλίματο και να περιορίσουμε την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας ε, στου λιγότερου από δύο βαθμού. Προσβλέπω τώρα στι δικέ σα απόψει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στους ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Εξ του ΕΛΚ, ο κύριος Γκάλερ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σαν εισηγητής για την έκθεση της Αρτικής, για τις δηλώσεις σας κύριε Επίτροπε, ιδιαίτερα για την εργασία της Επιτροπής όσον αφορά τις προτάσεις σας στους νέους στόχους για το 2020. Μας δείχνει πραγματικά ότι βρίσκομαστε στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων το θέμα της Αρκτικής και βεβαίως ε, με τις προτάσεις της εκθέσεις μου που είναι ρεαλιστικές, συγκεκριμένες, μας δείχνεται ότι ήδη είμαστε δεσμευμένοι. Δεν είναι τυχαίο το ότι σήμερα γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ. Στις 15 Μαΐου συναντώνται οι αρμόδιοι υπουργοί για το θέμα της Αττικής και εμείς είμαστε παρατηρητής σε αυτήν την συνάντηση. Θα ήθελα επίσης εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας, του ΕΛΚ, να εκφράσω αυτήν την σοβαρή δέσμευση. Βεβαίως και τα οικονομικά συμφέροντα σε αυτή την περιοχή είναι πολύ σημαντικά. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δεσμευθεί αρκετά. Η ανάπτυξη σε αυτή την περιοχή είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνουμε πολύ συγκεκριμένες ε, προτάσεις και βήματα έτσι ώστε να συνεχίσει η ανάπτυξη αυτής της περιοχής να γίνεται βάση βιώσιμων στόχων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ρυθμιστούν τομείς όπως η ναυσιπλοεία βάση του Διεθνούς Θαλάσσιου Δικαίου και άλλων φορέων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει συντονισμός στην πολιτική που αφορά την Αρκτική και η Ευρώπη με τα προγράμματά της, επενδύσεις της, την έρευνά της αλλά και την αγορά της να γίνει ένας πολύ σοβαρός εταίρος ο οποίος να συνεισφέρει σε αυτήν την αηφορία και την ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ισορροπημένοι όσον αφορά την πρόθεση διαφόρων συμφερόντων, κυρίως προωθώντας την αηφόρο ανάπτυξη. Επίσης, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, και αυτό είναι κάτι που το επαναλαμβάνουμε συνέχεια στους εταίρους μας προ το Βορρά, είναι πολύ σημαντικό κύριε Επίτροπε, ναι, να συνεχίσουμε την συζήτηση και το διάλογο για το θέμα της ενέργειας. Όμω, ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργό της Ισλανδίας έκανε κάποιες προτάσεις αναφέροντας το ενδιαφέρον που δείχνουν πολλές χώρες ασιατικές, η Κίνα. Δεν ανέφερε καθόλου την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν Ρώσοι, υπάρχουν ε, ε, Καναδοί, οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένη και επαγγελματική δραστηριότητα. Εμείς, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες συνεργασίας, οικονομικής συνεργασίας. Ναι, είμαστε ένας ε, παρατηρητής σε αυτές τις συναντήσεις, αλλά έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες. Δεν έχουμε εδώ μόνο τη δυνατότητα για διπλωματική δράση. Θα πρέπει πραγματικά να κινητοποιήσουμε τα δίκτυά μας και να κάνουμε μια πραγματικά οικονομική διπλωματία. Εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζουμε αυτή την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ για τους σοσιαλιστές. Παίρνει το λόγο κύριος, η κυρία Γιακονισάρη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις εισαγωγικέ σας παρατηρήσεις και για την αισιοδοξία που έχετε και για την πολιτική της Αρκτικής αλλά και για την ε, δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει το καστός μόνιμου παρατηρητή στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Βεβαίως, Καλό να μην γίνει η Αρκτική ένα Eldorado, όπως ε, πιστεύαμε τόσα χρόνια ότι θα αρχίσουν δηλαδή να τρέχουν όλα τα κράτη-μέλη για να βρουν ε, χρυσό και πρώτες ύλες. Και είναι πολύ δυσκολότερο να εξορυχθεί η πετρέλαιο από όσο νομίζαμε. Η ΣΕΛ, παραδείγματος χάρη, τα παράτησε γιατί είναι πολύ σκληρές οι συνθήκες. Αυτό είναι καλό γιατί τώρα έχουμε περισσότερο χρόνο από όσο νομίζαμε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την περιοχή με τρόπο ειρηνικό και βιώσιμο και να συμβαστούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων εκεί. Βεβαίω πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ της Αρκτικής και της Ανταρκτικής. Η Αρκτική δεν είναι μόνο το δεν είναι μόνο ο Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός, αλλά και κράτη που βρέχονται από αυτόν και λαοί που ζουν εκεί πέρα και βεβαίως ε, πρόκειται για την ε, πρώτη γενιά των αυτοχθόνων που πραγματικά λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντά τους. Εμένα μου πήρε συνέντευξη ένας ε, εκπρόσωπος των Σάμι στον βορρά στον αρκτικό κύκλο και με και ρώτησαν τι κάνει για μας η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει καν ότι υπάρχουμε και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά σε μας και είναι πολύ σημαντική ερώτηση και μία απάντηση σε αυτό είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Επίτροπος Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ίδρυση ενός κέντρου πληροφόρησης για την Αρκτική στο Ροβανιέμι. Και έτσι νομίζω θα μπορούσε να υπάρξει και μεγαλύτερη επαφή με τους ε, αυτόχθονες πληθυσμού. Και έτσι πραγματικά μπορούμε να δοκιθούμε σε μια ειρηνική εξέλιξη και να είμαστε καθυσυχασμένοι. Παραδείγματος χάρη η συνεργασία που υπάρχει, δηλαδή η Νορβηγία, παραδείγματος χάρη και η Ρωσία το 2010 συνεπέγραψαν μια συνθήκη και έτσι επιλύθηκαν διαφορές που είχαν για τη θάλασσα του Μπάρεντς. Και το Αρκτικό Συμβούλιο και η σημασία του έχει πραγματικά αυξημένο ρόλο και εκεί είναι το κατάλληλο πλαίσιο για να υπογράφονται συνθήκες. Επίσης, ε, οι υποδομές οι συγκοινωνιακές που δημιουργούνται ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενισχυθεί και η έκθεση του Κοινοβουλίου λέει πως είναι καλό να γίνουν αυτά από κοινού. Η βόρεια διάσταση θα μπορούσε να τα θέσει όλα αυτά υπό την αιγίδα της. Έχουμε λοιπόν όπως τόνισε ήδη και ο κύριος Γκάλερ, ο εισηγητής, ε, μεγάλη σημασία ε, που αποδίδεται στην πορεία αυτή διάσταση και χρειάζεται μια στρατηγική πολιτική, ειδικά όσον αφορά τις μεταφορές, ε, την επιμελητία και σημαντικό είναι να δούμε πώς θα συνδέσει η Κομισιόν την βόρεια διάσταση με την πολιτική για την Αρκτική. Και χρειαζόμαστε πιο λεπτομερή χρονοδιαγράμματα. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί, όπως είπαμε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτέλους έχει φτάσει η στιγμή για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και για αυτά για τα οποία είπατε για την έρευνα για αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι μπορούμε νομίζω να αιτιολογήσουμε την θέση του μόνιμου παρατηρητή που ζητάει στο Συμβούλιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις φιλελεύθερους. Κυρία Γέτνερ Μάκη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει πάγος, θάλασσα στην Αρκτική. Υπάρχουν όμως και 4 εκατομμύρια κάτοικοι, οι οποίοι θέλουν να αναπτυχθούν, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της περιοχής τους. Γι' αυτό και ακριβώς χρειαζόμαστε επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή της Αρκτικής. Δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να ξεχάσουμε και την βιοπικιλότητα. καθώς και την βιώσιμη ανάπτυξη των πόρων της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξη για την περιοχή της Αρκτικής. Γι' αυτό και η ομάδα μας στηρίζει την πρόταση να δημιουργηθεί μια τέτοια στρατηγική για την ανάπτυξη της Αρκτικής το συντομότερο δυνατόν. Αυτό θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και τους ε, αυτόχθονες λαούς τους κατοίκους δηλαδή της Αρκτικής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, διότι αναφέρατε την σημασία της δημιουργίας ενός κέντρου για την Αρκτική. Η ομάδα μας στηρίζει από την αρχή την ίδρυση ενός τέτοιου κέντρου πληροφοριών και πιστεύουμε ότι το πανεπιστήμιο το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει την σύνταξη μιας έκθεσης θα εισακουστεί και θα ιδρυθεί μια μέρα αυτό το κέντρο. Στηρίζω επίσης και τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει μόνιμος παρατηρητής στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Ο Επίτροπος ε, κατάλαβα ότι είναι υπέρ αυτής της ιδέας. Αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τους ε, κατοίκους αυτής της περιοχής τα θέματα που αφορούν την Αρκτική θα πρέπει να είναι προτεραιότητες στην ε, πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα θα μπει λίγο νωρίτερα στην ε, ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας και όχι τόσο αργά μέσα στη νύχτα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αντίστοιχη αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την περιοχή της Αρκτικής. Μήπως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε μια τέτοια αντιπροσωπεία, καθότι τα θέματα θα συζητηθούν πολύ καλύτερα από μια αντιπροσωπεία που θα έχει στο επίκεντρό της την Αρκτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Πρασίνων, ο κύριος Τάραν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εστονικά για να επιδείξω αλληλεγγύη με τους αυτόχθονες ε, πληθυσμούς της Αρκτικής. Το Μάρτιο του 2010 μπόρεσα να πάω στο ίδιο ε, εδώ, μάλλον συγγνώμη στην Ολομέλεια, μιλούσα για το ίδιο θέμα και τότε ε, ήταν η Κάθριν Άστον εδώ παρούσα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκανα έκκληση λοιπόν προς την κυρία Άστον να επιδείξει ιδεαλισμό και να προτείνει ένα μορατόριουμ για την εξόριξη των φυσικών πόρων της Αρκτικής. Βεβαίως είπα ότι εκπρόσωπος, όπως και αρκετοί συνάδελφοι εδώ στο Κοινοβούλιο, μου πρότειναν να είμαι λίγο πιο ρεαλιστής και για να είμαι ειλικρινής, δεν ε, φανταζόμουν ότι θα ήταν τόσο ιδεαλίστρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ε, ε ένιωσα την ανάγκη να το επισημάνω το γεγονό αυτό. Ε, από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε ρεαλισμό ούτε ιδεαλισμό επιδεικνύουν. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα 48 σημεία δράσης τα οποία προτάθηκαν το 2008. Δεν χρειάζεται κάποιο να είναι Βρετανό ευρωσκεπτικιστή για να γνωρίζει ότι κάθε φορά που υπάρχει πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει κάποιο νέο όργανο, είτε για... πρόκειται για την τραπεζική εποπτεία, είτε για οποιοδήποτε νομισματικό άλλο ζήτημα. Έχουμε καταφέρει όμως να κάνουμε κάτι για την Αρκτική. Υπάρχει προϋπολογισμός προς αυτό το σκοπό. Φυσικά και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να μειώσει και τη χρηματοδότηση στις επόμενες ε, πολιτικές προοπτικής ε, ε, κατά 12%. Εμείς θέλουμε να γίνουμε μόνιμοι παρατηρητές στο Αρκτικό Συμβούλιο, αλλά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν έχει ειδικού που να ασχολούνται με τη συγκεκριμένη πολιτική. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να λάβουμε θέση παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο, ενώ θα έπρεπε να προετοιμαστούμε, διότι διαφαίνεται όλο και περισσότερο ότι χρειαζόμαστε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και ο κόσμος χρειάζεται διεθνή διακυβέρνηση στην Αρκτική για να μπορέσει να το επιτύχει αυτό. Χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε βάσει ποιών προτύπων και με ποιο τρόπο θα γίνονται οι εξορίξεις, ε, με τι πόρους ε, συζητάμε και κατά πόσον θα χρησιμοποιηθούν στην Αρκτική ένοπλες δυνάμεις, ε, πώς θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες δυνατότητες για την εξέλιξη της Αρκτικής και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Ξέρω ότι η πλειονότητα των μελών του Κοινοβουλίου δεν είναι υπέρ της διακήρυξης της Αρκτικής ως ε, προστατευόμενη περιοχή. Να σας δώσω όμως ένα παράδειγμα από την Εστονία. Κάποιος ο οποίος μεγάλωσε στην Εστονία έδωσε το όνομά του σε ένα νησί στον Αρκτικό ωκεανό παρά το γεγονός ότι δεν πήγε ποτέ στην συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά 45 χρόνια αργότερα πήγε μια αποστολή που πρότεινε επίσης να ονομαστεί το νησί ε, στο όνομα του συγκεκριμένου Εστονού. Το 1976 δημιουργήθηκε το Συμβούλιο των Αυτοχθόνων Πληθυσμών και επιβεβαιώθηκε και ε, πέρσι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και αυτό το Συμβούλιο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν αυτά τα θέματα. Γιατί εμεί δεν κατανοούμε ότι χρειαζόμαστε να είμαστε και λίγο ιδεαλιστέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξ ονόματο ε, τη Ενωτική Αριστερά, ο κύριο Μέρφυ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη και πιο ιδιαστική απόδειξη της τρέλας του καπιταλισμού από την αντίδραση του κατεστημένων ανά τον κόσμο στο λιώσιμο των πάγων. Θα μπορούσε τα καλοκαίρια να μην έχει καθόλου πάγο σε 30 με 40 χρόνια. Η άνοδος λοιπόν της στάθμης της ε, θάλασσας και η ανάδραση του όλου φαινομένου θα έπρεπε να μας σοκάρουν. Ένα από τα χειρότερα σενάρια, εάν λιώσει και ο πάγος της Γρυλανδίας, θα μπορέσουν τα επίπεδα της θάλασσας κατά 7 μέτρα. Οπότε όχι μόνο το Μπαγκλαντές, αλλά και το Λονδίνο και το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη θα βρεθούν κάτω από το νερό. Αλλά αυτό το οποίο είναι εφιάλτης ε, για πολλούς ε, κάνει να τρέχουν τα σάλια στις εταιρείε ε, πετρελαίου. Άλλοι, μεταξύ των οποίων και η Κάθριν Άστον, καλωσορίζουν το άνοιγμα του βορείου διάβλου. Και αντιδρούν με έναν αγώνα δρόμου για την Αρκτική μεγάλη δυνάμει. Την επόμενη εβδομάδα οι περιβαλλοντικέ οργανώσει ζητούν μια παγκόσμια μέρα δράση για να στείλουν ένα μήνυμα κάτω τα χέρια από την Αρκτική. Για να φύγουμε από τη λογική τη ε, καπιταλιστική απληστία και να πάμε σε μια οικονομία χωρί ορυκτά καύσιμα. Κύριε Μέρφυ, δέχεστε μια μπλε κάρτα. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, πρώτα απ' όλα δέχεστε πως ο πληθυσμό που ζει εκεί έχει επίσης δικαίωμα στην ανάπτυξη και δεύτερον ε, σημειώνεται πως δεν τα έκαναν αυτά κάποιοι καπιταλιστές αλλά ένα κομμουνιστικό κινέζικο παγοθραυστικό έφτασε για πρώτη φορά ε, εκεί πέρα και ε, άνοιξε τον βόρειο θαλάσσιο διάβλο. Οι Κινέζοι κομμουνιστές θέλουν να τα κάνουν αυτά που λέτε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Βεβαίω, συμφωνώ. Τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών είναι, έχουν κορυφαία σημασία. Δεν νομίζω πως είναι υπέρ της καταστροφής του τόπου που ζούνε. Διαφωνούμε τώρα στο πώς ορίζουμε τις χώρες ως καπιταλιστικές ή κομμουνιστικές. Επειδή υπάρχει μια δικτατορία που αυτοαποκαλείται ε, κομμουνιστική, ε, δεν σημαίνει ε, πως είναι κιόλα. Υπάρχουν ε, διαφορετικέ ομάδε συμπεριελιστών, Κινέζων, ναι, Ρώσων, ναι, ε, Αμερικανών, ναι, Καναδών, ναι. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί και αυτή να μπει στο παιχνίδι. Στον εαυτό αγώνα για την Αρκτική. Και αυτοί που θα χάσουν θα είναι οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και ο πλανήτη μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στους επόμενους ομιλητέ. Η κυρία Εσάγια για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σε ένα μήνα το Αρκτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μόνιμος παρατηρητής ε, του Συμβουλίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναρωτιέμαστε αν πραγματικά μπορούμε να συνεισφέρουμε κάτι σε αυτή τη συνεργασία. Έχουμε κάποιους βιώσιμους στόχους για τη στρατηγική της Αρκτικής. Η ανακοίνωση του 2012 μας έδωσε βέβαια κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και θα ήθελα να σταθώ και στην προηγούμενη έκθεση του κυρίου Γκάλερ για την ε, βιώσιμη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρθηκε με πολύ σημαντικό τρόπο ο τουρισμός και κάποια άλλη κλάδοι που μπορούν να συνεισφέρουν ε, ε, στην περιοχή της Αρκτικής, αλλά ε, αναφέρθηκαν επίσης και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών. Καλό θα ήταν να υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο για την βιώσιμη και ευφυή ανάπτυξη της περιοχής και θα πρέπει να σκεφτούμε, όπως είπε και ο κύριος Φούλε, κατά πόσο θα πρέπει να συσταθεί αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ενημέρωσης για την Αρκτική. Ακούμε εδώ στην Ολομέλεια συζήτηση για αυτό το κέντρο στο Ροβανιέμι και το Ροβανιέμι σίγουρα θα μπορέσει να υποδεχθεί ε, το κέντρο αυτό για τη στρατηγική για την Αρκτική. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκάλαγκερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η προστασία και η διατήρηση της περιοχής της Αρκτικής σε αρμονικό τρόπο με τις επιδημίες του πληθυσμού της είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να γίνει στόχος. Πρέπει να στηρίξουμε και να προστατεύσουμε τις κοινότητες των αυτόχθων πληθυσμών. Σαφώς και θα πρέπει να μην ξεχνούμε τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων. Όπως ξέρετε πολλούν ε, ε, δέρμα φώκιας και πολλές φορές αυτό είναι και το μοναδικό τους εισόδημα. Ξέρετε πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μη γνωρίζοντα ε, τις συγκεκριμένες καταστάσεις αυτών των ανθρώπων βρίσκεται εκτός ε, αυτών των περιοχών. Σήμερα υπάρχουν εκπρόσωποι από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ισλανδία, τις βόρειες χώρες που είναι όχι παρατηρητές αλλά εμπλεκόμενα μέρη αυτής της ε, περιοχής και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει απλώς να γίνει ένας μόνιμος παρατηρωτής στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Χαιρετίζω αυτήν την ε, αίτηση που έκανε πολύ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει την παρουσία της στην Αρκτική. Δέχεστε μπλε κάρτα κύριε Γκάλαχερα. Αγαπητέ συνάδελφε, είπατε ότι οι αυτόχθονες λαοί έχουν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους σε κάποιες αποφάσεις στο παρελθόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πώληση δέρματος φώκιας. Ξέρετε ότι υπάρχει εξαίρεση για τις κοινότητες ε, που ζουν εκεί. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Στον τύπο στην, ε, στον Καναδά αυτή η εξαιρέση αναφέρεται πολλές φορές. Το γνωρίζετε. Όχι, δεν είναι αλήθεια στην πραγματικότητα και αυτό δεν είναι η άποψή μου. Είναι η άποψη αυτών που ζουν στη Γρυλανδία των αυτοχθόνων πραγματικά. Είναι η πραγματικότητα. Είναι γεγονός. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αν συναντηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους θα συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι υπάρχουν εκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια, πρέπει να περιμένουμε την τελική απόφαση, η οποία πιστεύω ότι θα έρθει σε λίγους μήνες. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό. Ο, συνάδελφος... Ο κύριος Άικχαουτ, σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, η στρατηγική της ε, Κομισιόν ε, με απογοήτευσε γιατί ακούω πράγματα όπως γνώση, ευθύνη, διάλογος και μιλάμε για ε, ε γεωτρήσεις χαμηλού κινδύνου. Τι εννοεί εδώ πέρα η Κομισιόν Ξεχνάτε το ότι η Κόνοκο Φίλιπς παραδείγματος χάρη αποφάσισε να μην προχωρήσει σε γεωτρήσεις το 2014 όπως λένε διάφορα ιδρύματα να μην ε, εξορίξουμε ποτέ τίποτα από αυτή την περιοχή η οποία πλήττεται δύο φορές περισσότερο από την ε, κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτή την περιοχή, να μην γίνουν ποτέ γεωτρήσεις εκεί πέρα. Και εσείς έρχεστε και μας μιλάτε για ε, γεωτρήσεις χαμηλού κινδύνου. Κούφια λόγια. Ευχαριστώ κύριο Πρέντα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο εισηγητής ε, για την Ισλανδία, ο υποφαινόμενος δηλαδή, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ε, ανάπτυξη της αρκτικής περιοχής. της Ισλανδία μπορεί να είναι μικρή χώρα, αλλά διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη περιοχή ε, είναι, έχουν τη γραμματεία του Αρκτικού Συμβουλίου, ο Ισλανδό είναι ο κάτοχο συγκεκριμένη θέση, Επομένω, είναι πολύ σημαντική η θέση τη Ισλανδία σε αυτό το πλαίσιο. Από την τελευταία συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ίδιο θέμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να εξετάζει τη δυνατότητα μια πολιτική ε, για την Αρκτική. Ε, και από εκεί και πέρα εξετάστηκαν ε, κατά πόσον υπάρχουν πολιτικές και διοικητικές δυνατότητες για κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι έχει φτάσει η στιγμή να αποφασίσουμε κατά πόσον θα έλουμε δική μας παρουσία στην περιοχή. Να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά στην έρευνα της περιοχής της Αρκτικής. Δόθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ στα τελευταία 4-5 χρόνια για την έρευνα στην συγκεκριμένη περιοχή. Εάν λοιπόν συμμετέχουμε ως μόνιμοι παρατηρητές στο Αρκτικό Συμβούλιο, θα αναλάβουμε φυσικά και τις ευθύνες μας. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να αναλάβουμε τέτοιον ρόλο εάν βρισκόμαστε εκτός. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα που έχουν πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για την ε, περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις κοινέ αξίες και αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών. Η Χώρε ε, τη Αρκτική και οι αυτόχθονε πληθυσμοί είναι αυτοί που έχουν τον τελευταίο λόγο, αλλά πρέπει και εμεί να συνεισφέρουμε. Ο κύριο Μπέλετ για 1,5 λεπτό. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ω ηγητή στην Επιτροπή Επιμηχανία, θα ήθελα να εστιαστώ στο συγκεκριμένο ζήτημα των ερευνών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αρκτική. Πράγματι, Υπήρξαν προσπάθειες της ΣΕΛ στην Αλάσκα που έδειξαν πως είναι πάρα πολύ δύσκολες οι επιχειρήσεις στην ε, Αρκτική και επικίνδυνες για τη φύση και την ανθρωπότητα. Πολλοί έχουν ζητήσει και εδώ μέσα ένα μορατόριο ε, των εξορίξεων στην Αρκτική. Όλοι γνωρίζουμε, πέρα από την ειδική περίπτωση βεβαίως της Γρυλανδίας, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ε, αρκτικά ύδατα. Όμως, το νέα σχεδιαζόμενη νομοθεσία για υπεράκτιες ε, ε, λειτουργίες πετρελαίου και αερίου υπάρχει μια σαφής υποχρέωση των εταιριών εξόριξης να αποδείξουν πώς μπορούν να αντιδράσουν αποτελεσματικά σε ατυχήματα και να περιορίσουν τις επιχειρήσεις τους όταν δεν μπορούν να αντιδράσουν. Μιλάμε για πραγματική υποχρέωση νομική και ισχύει αφορτιόρη σε πιθανές πλατφόρμες ε, στην Αρκτική. Βασιζόμαστε σε εσά λοιπόν κύριε Επίτροπε για να στηρίξετε αυτό το νομικό μέσο εντό του Συμβουλίου της Αρκτικής και ελπίζουμε ε, να είμαστε σύντομα εκεί μόνιμος παρατηρητής αλλά και στο διεθνές πλαίσιο με τους ε, βασικούς εμπλεκόμενους στο ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Ξυπ για 1,5 λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντική επιρροή στα τεκτενόμενα στην αρκτική περιοχή. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν σε αυτή την περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να γίνει μόνιμος παρατηρητής στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Πιστεύω ότι κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η δική μου χώρα ήδη είναι παρατηρητές και δεσμεύονται συμμετέχοντας ε, στα δρόμενα στην περιοχή αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν τα προγράμματα ανάπτυξης και πριν από λίγες, ε, λίγα χρόνια είχαμε μία έκθεση που αφορά ακριβώς την περιοχή της Αρκτικής, τον Βορρά. Κάποιες από τις τροπολογίες της έκθεσης αυτής δείχνουν ότι το ενδιαφέρον μας για την υποθαλάσσια περιοχή, για την εκμετάλλευση αυτών των περιοχών και των φυσικών πόρων είναι κάτι που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε πεπισμένοι ότι είναι πολύ σημαντική η διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοπικιλότητας ε, καθότι και η σταθεροποίηση του κλίματος, κάτι που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το τι θα κάνουμε σε αυτή την περιοχή. Οτιδήποτε λοιπόν κάνουμε θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε περίπτωση όπου θα εμφανιστεί κάποιος, θα βάλει μία σημαία σε μία περιοχή της Αρκτικής και θα θεωρήσει ότι είναι δική του περιοχή. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στη διαδικασία Κατσδιά. Η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Αρκτική είναι μια περιοχή στρατηγικής σημασίας και όλα είναι και περισσότερο αυξάνεται η σημασία της. το γεγονός ότι λιώνουν οι πάγοι βοήθησε να ανακαλυφθούν σημαντικά αποθέματα υδρογονανθράκων που ενδιαφέρουν φυσικά πολλές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιοχής. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική στρατηγική και να χρησιμοποιηθούν με κατάλληλο τρόπο οι πόροι της Αρκτικής. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος. Ε, οι ανεργειακοί πόροι που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή της Αρκτικής και θα ανακαλυφθούν στο μέλλον θα πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην πλήττονται τα οικοσυστήματα και επίσης ε, ε, με ανησυχεί το γεγονός ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για την εκμετάλλευση των πόρων της περιοχής. Ευχαριστώ ο κύριος Κάρας. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως την επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα έως Τετάρτη θα συνέλθει η κοινοβουλευτική διάσκεψη της Αρκτικής. Οπότε θα εκπροσωπήσω εκεί πέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα μεταφέρω τα όσα περιέχονται στο ψήφισμα, ειδικά την απέτηση το Αρκτικό Συμβούλιο του Μαΐου να εγκρίνει το καθεστώς παρατηρητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούω όμως πως έχουμε αντίρρηση του Καναδά και της Ρωσίας και παρακαλώ όλους τους παρόντες να χρησιμοποιήσουν όλες τις επαφές τους για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία του Μαΐου. Έχουμε τρία κράτη-μέλη που είναι πλήρη κράτη-μέλη, έχουμε έξι παρατηρητές, έχουμε την Ισλανδία που είναι υποψήφιο κράτος μέλος και έχουμε την κοινοβουλευτική διάσκεψη την επόμενη εβδομάδα για να χαράξουμε τη στρατηγική μας σε όλα αυτά τα θέματα και ζητάω και τη συνεργασία της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, Κύριε και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις σημαντικές συνεισφορές σας απόψε. Το Κοινοβούλιο αποτέλεσε κινητήρια δύναμη όσον αφορά την στρατηγική της Αρκτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και απόψε τονίσαμε για άλλη μια φορά πως ε, η Αρκτική είναι μια περιοχή που μας επηρεάζει όλους εδώ. Αναφέρθηκαν ε, επίσης ε, οι αυτόχθονες πληθυσμοί και να τονίσω ξεκάθαρα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει τους ε, κατάλληλους τρόπους για να διασφαλίσει τον ενημέρωση των αυτοχθόνων πληθυσμών για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχουν έναν τρόπο να εκφράσουν τις ανησυχίες τους στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα συνεχίσει τις διαδικασίες τακτικού διαλόγου με τους αυτόχρονους πληθυσμού. Ξεκαθαρίσατε πως η Αρκτική θα χρειαστεί στήριξη για να αντιμετωπίσει την, ε, τις τεράστιες οικονομικές και περιβαλλοντικές ε, προκλήσεις που είναι όχι μόνο σημερινές αλλά αφορούν και τις μελλοντικές γενιές. Η συνεργασία λοιπόν παίζει ένα ρόλο κλειδί και πρέπει να συνεισφέρουμε και εμείς και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα των γεωτρήσεων και εξόριξης ε, στην Αρκτική. Οι χώρες που βρέχονται από την Αρκτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κοινά συμφέροντα ε, για την σωστή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων που υπάρχουν στην ξηρά, τη θάλασσα και κάτω από τον πυθμένο της θάλασσας με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον και ωφελεί τις ε, τοπικές ε, κοινότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρέχεται από τον Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό οι περισσότερες γνωστές σήμερα πρώτες ύλες βρίσκονται εντός των ορίων της ζώνης των 200 μιλίων ή και εντός της υφαλοκρηπίδας των ε, κρατών που βρέχονται από το Βόρειο Παγωμένο Κένο. Επίσης, η συζήτηση εστίασε και στη συνεργασία με άλλες χώρες και ήδη εντείνουμε την συζήτηση με τις ΗΠΑ και τον Καναδά για την συνεργασία στην έρευνα στην Αρκτική. Έχουμε ένα τακτικό διάλογο με την Νορβηγία και ανταλλαγή απόψεων με την Ισλανδία για να βρεθούν οι δυνατότητες συνεργασίας. Επίσης έχουμε τις ε, δυνατότητες της ε, βόρειας ε, διάστασης. Η συνεργασία με την Καριλανδία θα δώσει νέες ευκαιρίες για να βοηθήσουμε. Τώρα η περαιτέρω εξέλιξη της πολιτικής βεβαίως εξαρτάται και θα εξαρτηθεί και από την πορεία της αίτησής μας στο Αρκτικό Συμβούλιο. Και θα ήθελα πριν απαντήσω στον ε, κύριο Κάρας να πω το εξή. Η στρατηγική της Αρκτικής όπως αναπτύσσεται στην ανακοίνωσή μας του 2012 δεν ε, είναι ακόμα μια πλήρης ανεπτυγμένη στρατηγική η πολιτική αυτή αναπτύσσεται από το 2008 και ακόμα βρίσκεται στην φάση της χάραξης οι συζητήσεις αυτές βοηθούν να οικοδομήσουμε και να βελτιώσουμε την πολιτική μας για να φτάσουμε κάποτε σε κάτι το οποίο θα είναι άξιο να λέγεται στρατηγική. Δηλαδή να έχουμε στενή συνεργασία μεταξύ της ΣΥΠΑ, της προσώπου αφενός και της ε, Κομισιόν χρησιμοποιώντας ε, όπως είπα όλους τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και διασφαλίζοντας την ε, συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Εν μεταξύ το έγγραφο εργασίας της ε, Κομισιόν ε, που κάνει μια απογραφή των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο χάραξης μιας ευρωπαϊκής αρκτικής πολιτικής αντιμετώπισαν τα περισσότερα από τα ζητήματα που έθιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικά όσον αφορά την ε, συνέπεια και συνεκτικότητα περιφερειακών και ερευνητικών προγραμμάτων και την ενίσχυση των επαφών με τους αυτόχθονες ε, πληθυσμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίες της επίσης συμμετέχουν ενεργά στο σύνομα εργασία ε, στις διάφορες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου της Αρκτικής. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ σύντομα στο θέμα της χρηματοδότησης ευκαιρίες ε, χρηματοδότησης ε, που υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή εξετάζονται στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος. Ο ορίζοντας 2020, περιφερειακά και διασυνοριακά προγράμματα πιθανότατα θα αποτελέσουν τομείς κλειδιά στο πλαίσιο της Ακτικής. Για να επανέλθω τώρα στην αίτησή μας ε, για το καθεστώς παρατηρητή. Ε, ευχαριστώ τον ε, βουλευτή, τον κύριο Κάρας. Ελπίζουμε τα μέλη του Συμβουλίου της Αρκτικής να καταλήξουν σε μια θετική απόφαση αναγνωρίζοντας τις σημαντικές συνεισφορές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να κάνει ακόμα στην πολύ σημαντική αυτή περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Η επόμενη συνεδρίαση αύριο, 5η 18 Απριλίου, από τις ε, 9 μέχρι τις 2 και από τις 3 μέχρι τις 5. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και έχει αναρτηθεί στο ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.